für alle ναι, τα χρηματιστήρια θα πρέπει να, να, γίνονται, να περνάνε από κεντρικό clearing και αυτό είναι σωστό. Μιλάμε για 146 ε, εταιρείε, επιχειρήσει, οι οποίε λένε ότι τα, οι δικέ μα λύσει, οι μεμονωμένε, δεν μπορούν να τυποποιούνται γιατί έτσι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να ε, παίξουμε στα χρηματιστήρια. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά και δύσκολα σημεία της νομοθεσίας που πρέπει να θέσουμε όρια μεταξύ των τυποποιημένων και μη τυποποιημένων, μεταξύ των απαιτήσεων για τα χρηματιστήρια και των απαιτήσεων για τις μεμονωμένες λύσεις που προτείνονται. Και αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε στα πλαίσια της ε, νομοθεσίας. Μετά μιλούμε για το επιχειρησιακό ρίσκο και την αξιολόγηση των, του, ρίσκου, του ρίσκου. Και το επόμενο σημείο είναι η αναγκαία διαφάνεια. Εκτός από μία γενική έτσι, εικόνα που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τις, ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Πληρωμές, δεν υπάρχουν πολύ σαφείς λεπτομέρειες για το τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και πριν και μετά την ε, εμπορική συναλλαγή. Αυτό προτείνει η Κομισιόν. Με αυτό λοιπόν το πακέτο, η Κομισιόν νομίζω έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο αντικατοπτρίζει και τις ε, προθέσεις του Κοινοβουλίου, δηλαδή να καλυφθούν όλα, όλοι οι τομείς σε ό,τι αφορά τα παράγωγα και εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που, προέκυψε και από το G20. Υπήρχαν και άλλοι τομείς οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα, αλλά στο, στην σύνοδο του G20 ε, αναφέρθηκε ότι πέρα από τη ρύθμιση των παραγώγων θέλουν ειδικά μέτρα έτσι ώστε να ε, να ε, αποφευθούν προβλήματα στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ε, τιμές των πρώτων υλών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σκόπιμο και απαραίτητο σε σχέση και με τις δικές μας υποχρεώσεις για την αγροτική παραγωγή και την παροχή τροφίμων ε, για όλους, ε, να μην εξαρτώμεθα από κερδοσκοπικά χρηματιστήρια και θα ήμουν ευγνώμων στην Κομισιόν εάν μπορούσε να κάνει δικέ τη προτάσει ή στα πλαίσια των ε, ρυθμίσεων για τα παράγωγα να εξεύρει μια λύση. Τελευταίο σημείο. Η αξιοπιστία τη αγορά και η εποπτεία δεν αφορούν μόνο τα παράγωγα, αλλά και άλλα προϊόντα, τα οποία ε, παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ στην νομοθεσία. Ε, ας πούμε πρέπει να αλλάξουμε τις αγορές για την κατάχρηση, τις οδηγίες για την κατάχρηση της αγοράς, πιστοποιητικά για το μέλλον, πώς θα είναι, στο, πώς θα είναι ο μορφότυπός τους. Εγώ προσπάθησα να δω τι γίνεται με την δημιουργία και την εκπόνηση των τιμών για τα, για τα προϊόντα ενέργειας και μετά υπάρχει και το αγαπημένο μας πρόγραμμα για, για τα πιστοποιητικά ενέργειας, για τα πιστοποιητικά εκπομπών. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Κομισιόν προτείνει η Εποπτική Αρχή στο μέλλον να έχει το δικαίωμα να περιορίζει τις θέσεις, δηλαδή υπό προϋποθέσεις, αν δηλαδή υπάρχει ε, καλυπτόμενο ίδιο κεφάλαιο, να ε, δώσει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές οι εμπλεκόμενοι στις αγορές να περιορίζονται. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σκόπιμο για τα, και για τα παράγωγα εντός χρηματιστηρίου θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος όγκος 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν χρειάζονται όμως ανώτατο όριο. Δεν χρειάζεται να θέσουμε ανώτατο όριο. Και ξέρω αρκετές με περιπτώσεις μεγάλων τραπεζών που ε, ο κίνδυνος τους φτάνει δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχουν λοιπόν ε, μεγάλες, ε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περιορισμούς εδώ, για όρια. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσουμε έγκαιρα εδώ στην Επιτροπή πριν από τις προτάσεις της Κομισιόν να κάνουμε μια έτσι, ενδελεχή ακρόαση. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Διαβάζω τους ομιλητές. Pascal Canvin, uh, Peter Skinner, uh, um, Και εγώ θα αφήσουμε κάπως να γίνει συζήτηση γιατί έχουμε αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την ψηφοφορία για τη φορολογία των συναλλαγών. Λοιπόν, έχουμε, έχετε το λόγο. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Λάγκεν για την εισαγωγή του. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα παράγωγα ως χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι πολύπλοκα και πολλές φορές ε, και, και χρησιμοποιούνται ε, οι προθεσμιακές συμβάσεις στα πλαίσια αυτά. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να διαφοροποιήσουμε τα προϊόντα ε, ανάλογα με την ικανότητά τους να δημιουργήσουν συστημικό κίνδυνο και την πολυπλοκότητά τους και να μην αντιμετωπίζουμε όλα τα συμβόλαια με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, θέλω να συγκεντρώσω τα σχόλιά μου σήμερα το πρωί σε του τελικού χρήστε. Επειδή ε, τι τελευταίε εβδομάδε ήρθα σε επαφή με του ψηφοφόρου μου και με πολλέ εταιρείε που χρησιμοποιούν τα παράγωγα αυτά ε, με ε, έναν τρόπο που να του ε, ε, καλύπτει στο δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο. Υπάρχουν ανησυχίε όσον αφορά τον την τυποποίηση και όλα αυτά τα οποία ανέφερε και ο υποψήφιο επίτροπο κ. Μπαρνιέ και σήμερα όπω ακούσαμε και από τον εισηγητή. Τα ζητήματα λοιπόν τα οποία αφορούν ε, την τυποποίηση και την αυξανόμενη ε, εγγύηση δημιουργούν ανησυχίες. Το 14% περίπου ε, των ε, συναλλαγών στα παράγωγα που προέρχονται από τους τελικούς ε, χρήστες θα καλύπτονται από τις εξαιρέσεις όσον αφορά τους κανόνες. Οι εταιρείε χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να μειώσουν τον κίνδυνο. Ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ορισμένους τομείς συμμετέχουν ενεργά στη χρησιμοποίηση των παραγώγων αυτών. Καταλαβαίνουμε βέβαια στους κινδύνους και το τι γίνεται με τη χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο δεν συμβάλλουν σε συστημικό κίνδυνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Γι' ζητώ ο εισηγητή και η Επιτροπή να ε, λάβουμε υπόψη ε, μια εξαίρεση για του τελικού χρήστε, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να μην αντιμετωπίζουν μειονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο όταν προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο του με τα παράγωγα. Ευχαριστώ. ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την τοποθέτηση του συναδέλφου του κυρίου Λάγκεν. Ε, θετική κρίση όσον αφορά την εργασία της Επιτροπής, χρησιμότητα της ε, χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, ανάγκη για να μην ε, τιμωρούνται αυτά τα προϊόντα χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, αλλά ταυτόχρονα και ανάγκη εισαγωγής μεγαλύτερης ρύθμισης, κυρίως όσον αφορά την αγορά των εξοχρημεστηριακών προϊόντων αυτών. Όπως είπε και ο κύριος Λάγκεν, το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι η αγορά φαίνεται ότι έχασε τον προσανατολισμό τη. Εγώ θα ήθελα και θα είμαι σύντομο, να αναφερθώ σε δύο σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τα εξετάσουμε σε ιδιαίτερο βάθος κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Το πρώτο σημείο αφορά τις ε, τις επιπτώσεις ε, ε, σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής αυτών των προϊόντων. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ανάγκη επαλήθευσης σε βάθος του εξή θέματο. Όταν δηλαδή η έλλειψη διαφάνεια ορισμένων από αυτών των προϊόντων έχει ω αποτέλεσμα τροποποίηση των φορολογικών εσόδων και οδηγεί σε φόρο διαφυγή. Νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το εξετάσουμε σε περισσότερο βάθο. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη χρήση των παραγόγων στη δημόσια διοίκηση, στα κράτη-μέλη. Και πιο συγκεκριμένα ε, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί πολύ συχνά κυρίως αν πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ε, μικρής διάστασης, δεν έχουν αυτοί οι οργανισμοί στη διάθεσή τους τα μέσα για να μπορέσουν να επαληθεύσουν τη βιωσιμότητα του προϊόντος που αγοράζουν. Ακριβώς για αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επαναδηλώσουμε την αρχή της ορθής παρουσίασης από λογιστική άποψη, κυρίως όσον αφορά τους δημόσιους συλλογισμούς αυτών των προϊόντων, προσφέροντας και αναφέροντας συγκεκριμένους κανόνες. Και γενικά πρέπει να πούμε ότι εδώ θα πρέπει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της έλλειψης διαφάνειας και να υποχρεώσουμε αυτούς που προσφέρουν ε, τέτοια προϊόντα κυρίως προς την τοπική αυτοδιοίκηση να εξηγούν ε, διεξοδικά το περιεχόμενό τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις επιπτώσεις τους, ε, τα αποτελέσματά τους, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ελπίζω λοιπόν είναι δυνατόν να μπορέσουμε ε, ε, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, εμεί ω Επιτροπή, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα προ το συμφέρον των πολιτών μα, αλλά και προ το συμφέρον τη εθνική διοίκηση σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ο Πασκάλ. Ευχαριστώ. Και η ομάδα μας εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις της Επιτροπής και για την ε, παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Λάγκεν των βασικών ε, διακυβευμάτων και ε, πρέπει να πω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την προσέγγιση του. Θα υποστηρίξουμε όλες τις προτάσεις που θα οδεύουν προς την έννοια της τυποποίησης των ε, προϊόντων τη μέγιστη τυποποίηση, συνειδητοποιώντα βέβαια απόλυτα ότι δεν μπορούμε να ε, φτάσουμε σε πλήρη τυποποίηση. Και προτεραιότητά μας επίσης θα είναι να διακρίνουμε σαφώς τα παράγωγα προϊόντα τα οποία οδηγούν σε συναλλαγέ ε, ε, που συνδέονται με την πραγματική οικονομία και σε, αυτού, και σε αυτά που αφορούν συναλλαγέ ε, σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση θέλει να εξασφαλιστεί έναντι του κινδύνου που συνδέεται με τη δική τη την οικονομική δραστηριότητα, τότε θεωρούμε ότι το παράγω προϊόν μπορεί να αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί επιτρέπει στην εταιρεία αυτή να ελαχιστοποιήσει του κινδύνου και να κάνει προγραμματισμό σε μεγαλύτερο επίπεδο από το βραχυπρόθεσμο επίπεδο τη αγορά. Αλλά σε πρώτο επίπεδο, η παρά, τα παράγωγα αυτά προϊόντα και η αγορά του είναι χρήσιμη για την πραγματική οικονομία. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μα, ε, δημιουργείται όταν τα δύο μέρη τη συναλλαγή είναι ε, ε, ε, είναι, ε, ε, δρούν σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο και δεν έχουν να κάνουν κάτι με την πραγματική αγορά, ισοτιμίε, ενέργεια κτλ. Εδώ βρισκόμαστε σε μια άλλη διάσταση, που κατά την άποψή μα είναι καθαρά κερδοσκοπική διάσταση. Γιατί δεν υπάρχει, αν θέλετε, οικονομικό συμφέρον στην αγορά. Δεν γίνεται δηλαδή προσπάθεια κάλυψη των κινδύνων, αλλά γίνεται προσπάθεια κερδοσκοπία μέσω τη ανάλυση των κινδύνων αυτών. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση και αυτή πρέπει να την, ε, ε, να την ε, περιορίσουμε συγκεκριμένα. Γιατί όπω είπε και ο κύριο Λάγκεν, μπαίνουμε σε μια λογική ατέρμονα. Και σε τελευταία ανάλυση, οι χρηματοπιστωτικέ ροέ εκρήγνεται γιατί, το ξαναλέω, δεν συνδέονται με την πραγματική οικονομία και μια πραγματική κάλυψη των οικονομικών κινδύνων. Αυτό λοιπόν αποτελεί τη βασική μα προσέγγιση όσον αφορά την έκθεση αυτή ε, και την, ε, και την ανάλυση των υφιστάμενων εργασιών και των μελλοντικών εργασιών της Επιτροπής. Το ξαναλέω, να διακρίνουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία ε, συνδέονται με τα παράγωγα και που οδηγούν σε πραγματική ασφάλεια και από την άλλη έχουμε μια απόλυτα χρηματοπιστωτική αντιμετώπιση και αυτό το απέδειξε και η κρίση, έτσι, ότι εάν δεν περιορίζεται με συγκεκριμένου κανόνες αυτή η δράση, τότε έχουμε συστημικούς κινδύνους και με δύο λόγια αδυναμία διαχείρισης αυτού του συστημικού κινδύνου κινδύνου εκ μέρου του επόπτη, συστημικού κινδύνου που προέρχεται από τα καθαρά χρηματοπιστωτικά ε, παράγωγα προϊόντα. Um, Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Διότι φαίνεται μεν σαν να είμαστε κατά όλων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που τελικά ως αποτέλεσμα τι θα υπάρξει, θα αναγκαστούν να υποστούν ορισμένους κανόνες που ίδιοι θα θεωρούν ότι βέβαια τους φλάπτουν. Ο κίνδυνος για μας είναι οι συνομιλητές μας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δηλαδή, να καταλήξουν να γίνουν ένα είδος μονοπωλίου με τυποποιημένα προϊόντα και γι' αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε τι ακριβώς, ποια ακριβώς από αυτά τα προϊόντα είναι ρεαλιστικά και λειτουργούν. Πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης και ο καταναλωτής σε τι στοχεύουμε, στην εξυπηρέτησή του. Δεν είμαστε απλώς εκφραστές ορισμένων ιδεολογιών ή απόψεων στην αγορά. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η κερδοσκοπία είναι κάτι το επικίνδυνο ναι, μπορεί να είναι επικίνδυνο, αλλά η ανάληψη κινδύνου γενικότερα δεν είναι αναγκαστικά κάτι αρνητικό. Πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ ανάληψης κινδύνου και κερδοσκοπίας. Δεν ταυτίζονται. Εάν τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, τότε μόνο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σαφή νομοθεσία, αντί απλώς να απαγορεύουμε ορισμένα πολύπλοκα προϊόντα απλώς γιατί είναι πιο εύκολο για μας διανοητικά. Αυτό που θέλουμε είναι το κατάλληλο επίπεδο νομοθεσίας να υπάρξει που να εξυπηρετεί και τον καταναλωτή και την βιομηχανία, λέει ο μιλητής, την τραπεζική βιομηχανία. Αρκεί τα κριτήρια να προέρχονται από την πραγματική οικονομία. Αν όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τραπεζίτες ορισμένα εργαλεία που διαθέτουν, τότε τους θέτουμε σε κίνδυνο πραγματικά. Ο κύριος Πορτάς. Εγώ έχω μια άλλη άποψη για τα παράγωγα προϊόντα από αυτήν που ακούσαμε προηγουμένως από τον τελευταίο μιλητή. Διότι από όσα ξέρουμε για τα προϊόντα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία της κρίσης που γνωρίζουμε. Απλώς ως λύση μετέφεραν το κόστος τους στον φορολογούμενο. Πρόκειται όμως για πρόβλημα που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Πρέπει βέβαια, έχει δίκιο ο συνάδελφος, να διαφοροποιήσουμε τα παράγωγα προϊόντα που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία και που στοχεύουν σε μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων, τα οποία προϊόντα είναι χρήσιμα και απαραίτητα, από τη μία και από την άλλη τις καθαρά κερδοσκοπικές δραστηριότητες επί των παραγόγων. Εγώ θα το έλεγα μάλιστα πιο ριζοσπαστικά από την Κομισιόν η οποία προτείνει απλώς κάποια νομική διευθέτηση. Εγώ νομίζω ότι καλό θα ήταν να απαγορευτούν πολλά από αυτά τα παράγωγα προϊόντα, να αποτιτλοποιηθούν. Ιδίως αν σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρισμού, τη γεωργία κτλ. Υπάρχουν πολλές προτάσεις που ακούστηκαν από την Επιτροπή πάντως. Η υποχρέωση κεντρικής αποζημίωσης, η υποχρεωτική κοινοποίηση όλων των δραστηριοτήτων και συναλλαγών και το μητρό τους. Νομίζω ότι αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά γιατί δημιουργούν μια πρόσθετη δυνατότητα που δεν την αναφέρει το κείμενο και που είναι η χρησιμοποίηση της φορολογικής ή δημοσιονομικής πολιτικής για ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση αυτών των παραγόγων προϊόντων. Με πληροφόρηση γίνεται αυτό, χωρίς όμως δεν γίνεται. Και κάτι άλλο ακόμη. Α, όχι κάτι άλλο, αυτά. η Βίκη, η Νίκη μάλλον. Σας κατευχαριστώ για τα, και για τα σχόλια που κάνατε ως προς το τι πρέπει να ξεκαθαριστεί και τι μπορεί να παραμείνει ως παράγωγο προϊόν θεμητό. Ως παράδειγμα είχα σκεφτεί κατά πόσον ο κύριος Γκόρζες δεν θα έπρεπε ορισμένες από τις τροπολογίες της δικής μας έκθεσης να τις αναλάβει εκείνος γιατί έτσι θα καταλάβαινε ποια είναι τυποποιημένα προϊόντα και ποια όχι. Ο κύριος Κορσές. Πρέπει νομίζω λοιπόν να δεχτούμε αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ των εκαθαριστικών οίκων και της κερδοσκοπίας και θα είναι και δικό τους συμφέρον να μειώσουν την ανάληψη κινδύνων από, για τη δημιουργία μεγαλύτερων πριμ. Θα ήταν καλύτερο να περιοριστεί ο αριθμός τους γιατί αλλά αυτό προϋποθέτει να γνωρίζουμε τι θέλουμε να καταργηθεί, πόσο κίνδυνο μπορεί να αναλάβει ένα σύστημα κλπ. Ο εισηγητής έθιξε ιδιαίτερα το θέμα των αγροτικών τιμών. Όπως γνωρίζετε η δική μου εκλογική περιφέρεια And, um, Η δική μου περιοχή λοιπόν είναι περιοχή παραγωγής σιτηρών και όλοι οι γεωργοί που γνωρίζω περιμένουν πρώτα να εκμεταλλευτούν στην αγορά για να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους πριν ψάξουν πολιτές. Και εδώ υπάρχει και μία σύνδεση με το πετρέλαιο γιατί χρησιμοποιούνται και παράγωγα του πετρελαίου στη γεωργία για λοιπάσματα κλπ. Κατανοούμε ότι υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις αγροτικές τιμές και ότι υπάρχει μια σύνδεση με την εξέλιξη άλλων τιμών εμπορευμάτων που συνδέονται όλα με το πετρέλαιο, αλλά τις διασυνδέσεις αυτές όπως μεταξύ γεωργικών προϊόντων και υπολείπων δημοσιονομικών αγορών δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε και δέχομαι την πρόσκληση, την έκκληση του εισηγητή για την οργάνωση ακροάσεως σχετικά. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα μιλήσω ως ε, σκιώδης από το ομάδα Άλντε. Θα συμφωνήσω με πολλά από όσα υπόθηκαν. Είναι σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των, ε, του κεντρικού clearing, αλλά όταν μιλούμε για κίνδυνο και για την χρηματοπιστωτική κρίση, δεν ήταν τα παράγωγα που δημιούργησαν την κρίση, αλλά μέσω της ε, κρίσης και κυρίως με την κατάρρευση της Lehman Brothers είδαμε ότι υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που είναι ανησυχητικά με όλες αυτές τις διαδικασίες που δεν μπορέσαν τελικά να κρατήσουν την, ε, τον ίδιο ρυθμό με ταχύτητα με την οποία μπορούν να απολυθούν τα παράγωγα. Αλλά αν είχε υποτιμηθεί ο κίνδυνος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να μην υπάρξει και υπερτίμηση του κινδύνου αν δηλαδή υπάρχει, μπορούμε να τιμολογήσουμε την, τον συστημικό κίνδυνο, θα πρέπει η τιμολόγηση αυτή να γίνει επί των συστημικών οργανισμών. Ας μην περάσει κατευθείαν στις ε, επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Πρέπει να δούμε βέβαια ποιος είναι στην άλλη άκρη από την, στη, τη σύναψη των συμφωνιών αυτών και πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά το υπάρχον κλίμα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανάταξη. Εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τα λογιστικά πρότυπα για να ορίσουμε ποιες είναι οι σωστές τραπεζικές μέθοδοι για το hedging και να δούμε τι γίνεται με το νόμιμο hedging και με το κερδοσκοπικό. Γιατί μπορεί να χρειάζεται όντως η υιοθέτηση τέτοιων προτύπων. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, τα σχόλια για την διαφάνεια είναι όλα α, θεμητά και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι να δω τι γίνεται με τον ανταγωνισμό και την διακριτική πρόσβαση σε φορείς clearing. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση. Θέλουμε ο κίνδυνος να ε, είναι συγκεντρωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα κατάχρησης της ιδιοκτησίας ή των υποδομών. Και όταν μιλούμε για την εποπτεία και τη διακυβέρνηση, επίσης είναι σημαντικό να, είναι, να υπάρχουν συνεκτικά α, πρότυπα. Ε, συνάδελφοι, εξακολουθούμε να συζητούμε, οπότε κάντε λίγο ησυχία αν θέλετε. Πριν την ψηφοφορία θα σας δώσουμε δύο-τρία λεπτά για να συζητήσετε αυτά που συζητάτε τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει και ομάδα εργασίας για τα παραγωγά με το στο Συμβούλιο και Ούτως ή άλλως η θέση του Κοινοβουλίου είναι σημαντική ως συνομοθέτη, οπότε νομίζω ότι η Κομισιόν πρέπει τώρα να πάρει το λόγο για να μας απαντήσει και αν θέλεις Πάτρικ να είσαι σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Τέσσερις παρατηρήσεις θα κάνω πιστεύω ότι σχεδόν όλα όσα λέχθησαν σήμερα είναι σχετικά και σημαντικά. Τα παράγωγα είναι χρήσιμα, είναι ζωτική σημασία στην οικονομία μα, για τι επιχειρήσει μα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που, ε, που έχουν μπροστά του. Κανεί δεν διαφωνεί. Τα παράγωγα δεν προκάλεσαν την κρίση, αυτή την κρίση. Το ξαναλέω, τα παράγωγα δεν προκάλεσαν αυτή την κρίση, αλλά συγκέντρωσαν τον κίνδυνο και απέκρυψαν τον κίνδυνο του χρηματοπιστωτικού μα συστήματο τα παράγωγα είναι παγκόσμια προϊόντα, δρούν σε παγκόσμια αγορά, άρα χρειαζόμαστε και παγκόσμιε συνολικέ λύσει. Δεν μπορούμε εμεί μόνο στην Ευρώπη να βρούμε λύσει ε, οι οποίε δεν θα ευσταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει συμφωνία ε, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο για τη ρύθμιση και το είπε και ο Επίτροπο Μαγκρίβη. Θέλουμε μια, σημαντική στάση και συνολική. Πρέπει να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό και πρέπει να κάνουμε μια βασική στροφή. Αλλά η νομοθεσία μα και η ρύθμισή μα να είναι λογική ε, και χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πώς το κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία ακόμα και σε μεγάλο μέρο τη τραπεζική κοινότητα. Όχι σε όλου, αλλά οι περισσότεροι από του ίδιου τραπεζίτε υποστηρίζουν την ανάγκη για ε, κεντρικό συμψηφισμό, ο οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά και απομακρύνει τον κίνδυνο από το σύστημα. Αλλά πρέπει να είμαστε σαφεί ότι δεν μπορούμε να ε, δρούμε όλοι σε κεντρικό επίπεδο. Δεν μπορούν όλα τα τυποποιημένα προϊόντα να αποτελούν αντικείμενο συμψηφισμού σε κεντρικό επίπεδο και να αποτελούν αντικείμενο τυποποίηση. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε σωστά και να μην υπάρχει παρεξήγηση γύρω από το τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο τυποποίηση και τι όχι. Και εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε διμερεί συμβόλαια παραγόγων που να μην είναι τυποποιημένα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο τη επιχειρήσει. Επόμενη παρατήρηση. Τελικοί χρήστε. Πάρα πολύ σημαντικό. Εταιρικοί τελικοί χρήστε που χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να διαχειριστούν τον κίνδυνό του. Από το 1991 το πράττουν και θα εξακολουθήσουν να το πράττουν. Αλλά σε τελευταία ανάλυση οι τελικοί χρήστες ή ε, οι εταιρείε ε, ε, προχώρησαν στη σύναψη συμβολέων που δεν είχαν τιμολογηθεί κάτω από ό,τι θα έπρεπε. Και άρα παρασύρθηκαν στα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η χρηματοπιστωτική κρίση. Άρα οι εταιρικοί τελικοί χρήστε έμεσα είναι μέρο του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Πώ λοιπόν πρέπει να του αντιμετωπίσουμε. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί εταιρικοί τελικοί χρήστες ε, που από συστημική άποψη είναι ε, σημαντικοί γιατί σε αυτούς πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, τους συστημικά σημαντικούς. Ναι, και εκεί να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα και τι κινδύνους πρέπει να δούμε. Οι υπόλοιποι προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα λογικό τρόπο για να μπορούν να εξακολουθούν να διαχειρίζονται το κίνδυνό τους και να δρουν θετικά στην οικονομία. Δεύτερη παρατήρηση, τρίτη παρατήρηση μάλλον ότι ε, όλοι αυτοί ε, ε, συνάπτουν συμβόλαια μέσω μεσολαβητών, μέσω τραπεζών, που θα πρέπει να αξιολογούν και να τιμολογούν τον κίνδυνο σωστά. Επανεξετάζουν οι τραπεζίτες αυτό το θέμα, γιατί σε τελευταία ανάλυση ο κίνδυνος αυτός περνάει στους τελικούς χρήστες. Είτε ρυθμίζονται τα παράγωγα σε κεντρικό επίπεδο, είτε όχι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πιο ρεαλιστικές τιμές για τις συμφωνίες αυτές. Και επόμενη παρατήρηση. Προφανώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα είμαι σύντομος, αλλά αν κινηθούμε ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση του κεντρικού συμψηφισμού και δεν ε, συνδέσουμε αυτόν τον κεντρικό συμψηφισμό με αυστηρέ ρυθμίσει, ε, φτιάχνουμε τα θεμέλια για την επόμενη κρίση. Θέλουμε υψηλότερα ε, πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι αυτούς ε, αυτά τα εμβαλωματικά μέτρα και αυτού του ε, σποραδικού κανόνε. Και πρέπει να δούμε και το θέμα τη πρόσβαση στην αγορά. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα όπου με βάση τα υφιστάμενα 10 γραφεία του συμψηφισμού, γραφεία συμψηφισμού είναι μονοπόλια. Θέλουμε ε, λειτουργησιμότητα, να δούμε το θέμα ε, της, ε, ε, ε της υποβολής έκθεσης όσον αφορά τη θέση. Θα έρθουμε σε επαφή με τους συνάδελφους Γεωργίας. Επίση, ε, Ιούνιο-Ιούλιο ε, έχει δεσμευτεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ο κ. Μπαρνιέ. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, τεχνικές, έχει επιτροπές σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων και όχι, σε, και όχι του Συμβουλίου, για να δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Και θέλουμε ε, να, σα να σας ζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ε, κατά πόσο θα συμφωνήσατε να κάνουμε εργαστήρια με τα μέλη τη Επιτροπή για το θέμα αυτό για να ανταλλάξουμε απόψει σε θέματα κοινού ενδιαφέροντο. Σα ευχαριστώ για αυτή την προσφορά. Θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ακολουθήσουμε την προσφορά σας. Τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να ε, κλείσει το θέμα. Ε, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις τους. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν αυτό που είπα και εγώ στην αρχική μου παρέμβαση. Ίσως η ε, προσέγγιση να ήταν λίγο διαφορετική, αλλά είναι σαφές ότι αυτές, αυτοί οι κεντρικοί οργανισμοί συμψηφισμών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να μην είναι δημιουργημένοι από τις αγορές, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για όλα τα παραγωγικά προϊόντα. Δεύτερον, φυσικά υπάρχουν και διμερείς συμβάσεις, συμφωνίες και το θέμα είναι πώς μπορούμε να επιτύχουμε τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα εκτός χρηματιστηρίου χωρίς συμψηφισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά μόνο όταν έχουν μεγαλύτερο, ε, μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν μικρότερο κίνδυνο από ότι αν, αν είχαν υποστεί συμψηφισμό για τις, ε, για τις μεταρρυθμίσεις. Ε, πόσο ξέρω η Κομισιόν για τα διμερεί παράγωγα θέλει να, εκδώσει, να προτείνει για τις ε, υψηλότερες τιμές για τις τράπεζες. Ε, όλο αυτό λοιπόν το θέμα ε, συνδέεται και με τις υπόλοιπες διατάξεις και σε αντίθεση με, την, ε, με τους υπαλλήλους της Κομισιόν που γενικώ συμμερίζουμε τις απόψεις τους αλλά για, αυτή την, για κάθε μεμονωμένη διάταξη έρχεται πάντα η απάντηση ναι αλλά δεν έφυγε αυτός ο τομέας για την κρίση ε, εντάξει αλλά δεν μπορούμε να, κάνουμε τέτοιες, να κάνουμε πολιτική με τέτοιες απόψεις. Φυσικά δεν είναι απλά τα πράγματα και δείτε και τον πίνακα, ο όγκος των παραγόγων εκτός χρηματιστηρίων τον Ιούνιο του 2008 ήταν 683 δισεκατομμύρια δολάρια. 458 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν ε, φόροι. Ε, προς όλες τις ε, δυνατότητες, κερδοσκοπία, και ε, κτλ. Μετά, επιστοτικές συμβάσεις 75 δισεκατομμύρια και απόλυτα ανασφαλή 81,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε φυσικά υπήρξε κερδοσκοπία, φυσικά ε, κερδίθηκαν πολλά χρήματα μέσω το, της δημιουργίας παραγόγων που εστάλησαν στην αγορά και δεν υπήρξε καμία εξασφάλιση ό,τι αφορά το ρίσκο. τα βραχυπρόθεσμα κέρδη αποταμιεύθηκαν. Ας δείτε, δείτε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Με, το νέο, με τα νέα κέρδη που έχει η Goldman Sachs. 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι λοιπόν αξιόλογο το πώς, ε, πώς συμβαίνει αυτό. Ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι ο δικός μου ο τομέας δεν φταίει για την κρίση. Ε, πάντα οι άλλοι φταίνε, το ξέρω αυτό. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι ε, η, όλη αυτή η διαδικασία με την αποτυχία της, των αγορών παραγόγων έχει να κάνει και με την διαχείρισή τους από τις τράπεζες. Φυσικά έχει συμβάλει και αυτό στην ε, κρίση. Ελπίζω η Κομισιό να μα δώσει ε, σύντομα πληροφορίε, να δούμε τι γίνεται και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Νομίζω ότι και αυτό κινείται προ σωστή κατεύθυνση. Και ε, ελπίσουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να οργανώσουμε μία ακρόαση εδώ στο Κοινοβούλιο. Εντάξει, τα εργαστήρια είναι καλά, ωραία, μπορούμε να λειτουργήσουμε πολύ καλά στι τεχνικέ προδιαγραφέ, αλλά άλλο είναι το, η δημόσια ακρόαση του Κοινοβουλίου που πρέπει να αποτελεί την ανοιχτή σκηνή διαβούλευση. Οπότε, Πρόεδρε, ε, ίσως το Μάη, αν μπορείτε, ε, ή τέλος ε, Απριλίου, ας ε, οργανώσουμε μια μεγάλη δημόσια ακρόαση με συμμετοχή των εμπορευομένων, των αγορών, εδώ στο Κοινοβούλιο. Και εγώ, στην έκθεσή μου, το αναφέρω αυτό, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι βέβαια, θα σας το υποβάλω, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα για πρώτη φορά συζητούμε το θέμα αυτό. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank, you very much. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα είναι ως εξής. Η έκθεση θα εξεταστεί στις 22 Φεβρουαρίου. Προσωρινά η προθεσμία της τροπολογίας, λοιπόν, είναι η 1η Μαρτίου. Και βεβαίως θα επαναξετάσουμε την ημερομηνία αυτή στις 22. Ε, Ίσως θα πρέπει να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να έχουμε και μία ακρόαση. Πάντω θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε την ψηφορία μα έγκαιρα για, την, για να μπορέσει ε, να είναι και χρήσιμη η έκθεση αυτή στην Επιτροπή. Λοιπόν, τέλο πάντων, τελειώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και τώρα θα πάμε στι ψηφορίε. Όλοι λοιπόν, εξ από έχουν τον, έχετε, ε, οι υπόλοιποι έχετε πάρει τον κατάλογο ψηφοφορίας. Right. As we, as we move to the... Ωραία. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Δεν κάνετε και λίγο ησυχία, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να μην ακούσετε τις ανακοινώσεις. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των ομάδων για να αναβάλουμε την ψηφορία για, για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα ε, ξεκάθαρε οι ομάδε για τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Είπαμε λοιπόν καλύτερα να, το, ε, να είμαστε ε, καλυμμένοι παρά να βιαστούμε. Δεύτερον, σα ζητήσαμε να φέρετε τι κάρτε σα. Για να δούμε, επειδή έχουμε και πολλά έξτρα μέλη και μπορεί κατά καταμέτρηση να είναι δύσκολη. Για να δούμε λοιπόν, για βγάλετε τις κάρτες σας. Just search for mine. ok. Bonjour. Merci. Merci. Merci. Ça va. Everything is... Okay. Right, that's my card. Jean-Paul. Right. Est-ce que tu seras aujourd'hui... No, it's in... Sorry, is anybody in difficulty? Κάποιος δεν έχει κάρτα σοφορίας. Είστε όλοι εντάξει. Ωραία. Αν πρέπει να μετρήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα. Ωραία. Ο κύριος Κάρας δεν έχει κάρτα. Ο κύριος Γκίγκελ. A lot oh, <laughs> um, yeah, okay. Right, the, the Ωραία. Πρώτη ψηφοφορία. Έκθεση της κυρίας Αλβάρες. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Είμαστε έτοιμοι. Θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε με ανάταση των χεριών και μόνο αν δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω τον συμβασμό Α. Υπέρ. Ε κατά αποχές εγκρίθηκε. Οπότε πάμε στην τροπολογία 8. Τροπολογία 8. Εισηγητή υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11, τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 12, τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχουμε τώρα το συμβασμό B, το Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε πάμε τώρα στη 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13, τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 14. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Δεν δουλεύει. Το δικό μου δεν δουλεύει.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 Νομίζω ότι... Διακόπτη πρόεδρος. Ωραία. Δεν σηκώνουμε τα χέρια γιατί να παίζουμε με τα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Λέει η Well, okay. Ε, we all know that we have to leave our voting cards in. Λοιπόν, αφού έχουν οι περισσότεροι τις κάρτες τους, εκτός αν μερικοί τι βγήκε 20 υπέρ λέει και 21 κατά Μια στιγμή κύριε έχετε τώρα κάρτα. Πρόεδρε, βλέπω ότι δεν λειτουργεί η κάρτα του κυρίου Σικλούνα, ενώ την έχει βάλει μέσα στο, στο μηχάνημα. Μάλλον πρέπει να το μετρήσετε έτσι, με το χέρι το δικό του, τη δική του την ψήφο. Κύριε Κάρας, εσάς δουλεύει η κάρτα σας. Ωραία. Ε, τότε ο μόνος που έχει πρόβλημα είναι ο κύριος Σικλούνα και ο κύριος Σάιμον. Ψηφίζουν υπέρ. Το μετράμε και αυτό. 22 λοιπόν υπέρ και 21 ψήφι κατά. Όχι δεν γίνονται αυτά κραυγές. Πρόεδρε, ε, δεν είναι μαθηματική άσκηση τώρα εδώ πέρα. Α ψηφίσουμε δια ανάταση τη χειρό. Α μετρήσουμε, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό που κάνετε. Μισά με το χέρι και μισά με το μηχάνημα. Ε, Μα αυτό φταίει το μηχάνημα, δεν φταίνει οι βουλευτέ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μετρηθούν όλες οι ψήφοι. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει η μεικτή μέθοδος, τότε θα κάνουμε διανατάσεως της χειρός. Okay. Ωραία. Hang on. We, we now have a Περιμένετε. Λοιπόν, ο κύριος Σικλούνα στο μηχάνημά του τώρα δουλεύει και το μόνο που δεν δουλεύει είναι του κύριου Σίμων. Λοιπόν, γιατί να μην ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα. Γνωρίζουμε ότι πάντα πρέπει να μετράμε και έναν με το χέρι. Λοιπόν, ψηφίστε λοιπόν τώρα ηλεκτρονικά για την τροπολογία 14. 14. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Λίγη η ψηφοφορία. Αμάν. Κι άλλος. Κοιτάξτε. Φαίνεται ότι... Πώς δούλεψε. Α, δούλεψε. Έληξε η ψηφοφορία, είπα. Δεν μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε. Λοιπόν, θα το ξανακάνουμε διανατάσεως. Διανατάσεως. Ε, αντί να κάνω, άμα δεν δουλεύει η μηχανή, λοιπόν, υπέρ διανατάσεως. 21 υπέρ. Κατά. Τα. Α, φαίνεται τώρα είναι περισσότεροι ψήφοι κατά 24 ή 25. Άρα μάλλον έχει απορριφθεί. Καμία αποχή. Όχι. Εντάξει. Ωραία. Η 14 απερίφθη. Τώρα η 38 υπέρ διανατάσεως. Τα αποχές εγκρίνεται. Η 15 αποσύρε, έχει αποσυρθεί. Για την 39 τώρα. Υπέρ της 39, υπέρ. Κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αν θέλετε μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ. Όχι, ξανά με τα χέρια. Υπέρ. Υπέρ. Ναι, είπα ξανά. Υπέρ, ξανά, υπέρ. Για την 39, υπέρ. 39. Παρακαλώ να έχετε τα χέρια ψηλά γιατί μετράμε. Δεκαοχτώ μάλλον. Κατά. 20 αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η 16 υπέρ Όχι, κοιτάξτε, Ψηφίσαμε. Αν μερικοί δεν σηκώσουν το χέρι δεν μετρούνται. Λοιπόν, 16 είπα. Όχι, εγώ μέτρησα αλλιώ. Δεν ήταν. Όχι, έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 16 υπέρ. 16 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές ξανά υπέρ Ξανά Πρέπει να βάλουμε ψηφολέκτες, δεν γίνεται. Ψηλά τα χέρια παρακαλώ. 22. Μην ανακατεύεσαι συνέχεια, Βέρνερ. Η γραμματεία μέτρησε 22 υπέρ. Κατά Νομίζω ότι για πιο γρήγορη ψηφοφορία, για έλεγχο, ο συνάδελφός μου εδώ δεν θα ψηφίσει και μπορούμε να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Καλά, ας το δοκιμάσουμε ηλεκτρονικά τώρα. Ή μάλλον εγώ δεν θα ψηφίσω και ο συνάδελφός μου θα ψηφίσει. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ποια τροπολογία? Ένα, τροπολογία ένα, ηλεκτρονικός έλεγχος και επαλήθευση. Έληξε υπέρ 22 κατά 24. Ωραία. Απορρίπτεται. Και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία δουλεύει. Λοιπόν, τώρα η τροπολογία 2 υπέρ. Γιατί όχι ηλεκτρονικά, αν Ναι, μπορούμε και ηλεκτρονικά λοιπόν. Αλλά αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Η Ιωάννη Παύλε ψηφίζει. Λοιπόν, ψήφισαν όλοι. Έληξε. 22 υπέρ 23 ε, κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα η τρία. Ας την κάνουμε και αυτήν ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τρία. Είναι ένας παραπάνω. Α, Ένας παραπάνω από το έλκυνε. Ποιος δεν θα ψηφίσει παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει τώρα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, λίγη ψηφοφορία, 23 υπέρ 22 κατά. Εγκρίνεται 17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 Ας ψηφίσουμε τώρα για το κείμενο ή ηλεκτρονικά, όπως ε, τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 5 κατά και 4 αποχές. Ας κάνουμε το ίδιο και για το νομοθετικό ψήφισμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Έχετε ψηφίσει όλοι. Έχουμε τους σωστούς ψηφίζοντες. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 4 κατά και 4 αποχές. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Συγχαρητήρια στην ε, Εισηγητρία. Πάμε στην αμοιβαία συνδρομή για την ίσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. Έτοιμοι. Τροπολογία 2. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είναι σαφές αν απέχετε. κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Απέχετε. Δεν είσαστε κατά. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ για την τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στον συμβαστικό, συμβαστική πρόταση α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Νομίζω τώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. It Okay. everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Ακόμα περιμένουμε να μας πει ο πίνακας τι έγινε με την ψηφοφορία. 41 υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Πάμε για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το νομοθετικό ψήφισμα. I don't understand why it takes so long for the numbers to stabilise, but it... Um, is it, is it, it's a vote... Right, the vote is closed. Πέρας Θα τον προσθέσουμε τον Σάιμον, εντάξει. 38 υπέρ, 0 ψήφι κατά και μία αποχή. Αλλά θα προσθέσουμε και μία. Για το, γιατί ο ψηφίζων εξ ονόματος του κυρίου Σάιμον έχει φύγει. Ε, εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Nine. And now we vote on item 10. Πάμε στο 10. Προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης. Ready? The... Somebody said no. Is everybody ready? Είστε έτοιμοι όλοι? Okay. Amendment 5. Τροποποίηση, τροπολογία, συγγνώμη, 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική πρόταση α υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά αυτό. Την τροπολογία 18 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Um, is... Have any problem? You will count Υπάρχει πρόβλημα. It's okay? Yeah. All right. Okay. So those in favor? Yeah, Mr. Simon, we have to add in again. Mrs. Θα προσθέσουμε τον κύριο Σίμων και πάλι. Πέρας ψηφοφορίας. 20 Υπέρ 23 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. Ε, το... Ε, συμβαστική πρόταση B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. 23. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά και αυτό. Τροπολογία 23. Okay, yeah. Has everybody voted? Right, Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Την προσπέρασα μία. Πάμε λίγο. Πάμε στη 2. Τροπολογία δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ή. E. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφός επί της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Has everybody voted? Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Okay. Well, we'll close the vote. Okay, yeah. So that is 43 in favor and one abstention, including... 43 υπέρ, μία αποχή. Ε, ψηφίζουμε επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Vote is closed. And that's the same, 43 υπέρ και μία ψήφος κατά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε στο σημείο 11. Έκθεση του κυρίου Ντομενίτσι για την προαιώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα. Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, συμβαστική πρόταση α. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Την 25. Πάμε στην παράγραφο 3. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά για να είμαστε σίγουροι. Για την 28. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 28. Votes closed. περασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22-19. Πάμε στον συμβαστική πρόταση B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω θα το ελέγξουμε και αυτό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 33. Vote is closed. And that is carried. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Τροπολογία 36 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι ήταν σαφές, αλλά εντάξει, αφού θέλετε ας το ελέγξουμε. 36. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σας το είπα. Απορρίπτεται, το είπαμε, απορρίπτεται. 35. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται.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 Ξανά, ξανά. Δεν μπορούμε να, την, ξαναψηφίσουμε επειδή κάποιο μπήκε τώρα. Ψηφίσαμε. Ναι, αλλά δεν δουλεύει το μηχάνημα του κυρίου Σίμων. 21, εγκρίνεται είπαμε. 38, υπέρ. Τροπολογία 38, υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε. Τροπολογία 38. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. is closed. Oh, no, it's not closed, Mr. Right. It does. Okay, so... Ωραία. Θα προσθέσουμε ένα σοσιαλιστή. Εγκρίνεται λοιπόν. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση Ή. Υπέρ. Συμβιβαστική πρόταση Ή. Υπέρ. Ε, κάνετε πολύ φασαρία όμως. Συμβιβαστική πρόταση Ή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Για να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 40. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. 23 με 20. Πάμε στην παράγραφο 10, αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στο συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, ε, εκτιμώντας 1 ως 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, Κατά. Αποχές. Λυπάμαι, πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Right, we all voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 22 με 19. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω το ίδιο. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο. Εκτιμώντας 5 και 6. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 3. περας πληροφορια ψηφοφορίας. Καταπίπτει. 21-21, άρα απορρίπτεται. Απορρίπτεται, δεν καταπίπτει, απορρίπτεται. ε, 7 7-20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική M, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω καλό θα ήταν να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5 ηλεκτρονικά. Right, vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Μπερδεύτηκα τώρα. Το ΕΛΚ τι ακριβώς κάνει. Right, if you, if you can't put your hands up, we'll have to do it. Αν δεν μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας, πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Α, λοιπόν, ε, ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 6. What am I doing? Okay, the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επτά. Υπέρ. Υπέρ για την επτά. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε και αυτό. Τροπολογία Έπτα. Has everybody voted? Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Ο κύριος Σίμων προστίθεται στους υπερψηφίσαντες. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Μία κάρτα εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Συμβαστική N. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Κανένα δεν σηκώνει το χέρι του. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 9. Κατά. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προσθέτουμε και τον κύριο Σίμων. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική O. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 12. Vote περας πληροφοριας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23-20. Τροπολογία 14. Υπέρ. Ε, ο, ε, εκτιμώντας δέλτα, ε, αρχικό κείμενο. Αρχικό κείμενο, το ξέχασα αυτό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 τώρα. Υπέρ κατά αποχές. Τι θα γίνει με τα χέρια σας, πάλι πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σας, οπότε και εγώ πώς να ξέρω. There we go. My vote's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22-21. Τροπολογία 16. Κάντε λίγο ησυχία. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 19, η οποία δεν καταπίπτει. Τροπολογία 19, λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Votes closed. Oh. Πέρας ψηφοφορίας. Σχεδόν πέρας ψηφοφορίας. Τώρα πέρας ψηφοφορίας. Πρόεδρε, το κούρασες. Μια πρόταση δεν μπορεί να κάνει αυτή η γυναίκα. Εγκρίνεται το, η έκθεση. Πάμε στο σημείο 12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2008. Okay, all right, okay. Okay, so we now vote on paragraph... Πάμε στην παράγραφο 1. Jean-Paul. Ε, Ήθελα να πω ε, το εξή του συναδέλφου του ΕΛΚ, ότι υπήρξε μία τροπολογία όσον αφορά τον κατάλογο ψηφοφορία. Ψηφίζουμε θετικά για την τροπολογία 59 και θετικά και ε, για την 69. Έτσι. Να σα πω και το εξή. Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, νομίζω ότι όσον αφορά τις τροπολογίες του IFM θα πρέπει να προβλέψουμε δύο ημέρες ψηφοφορίας. Έτσι το λέω, για γελάσουμε και λίγο. Ζαν ε, Jean Paul, upon you to get. Jean Paul, στηριζόμαστε σε σένα για να έχουμε πολλούς συμβιβασμούς. Λοιπόν, παράγραφος 1. Υπέρ, κατά, αποχές, πέρασε. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, δεν σηκώθηκαν αρκετά χέρια. Θα ελέγξουμε. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Πέρασε. Παράγραφος 2. Τροπολογία 12. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά αποχές, περνάει. 14 υπέρ, κατά, πρέπει να ελέγξουμε. Άρχη του ψηφοφορία στη 14. Ψηφίσατε. Έκλεισε. Πέρασε σαφώ. Παράγραφος 4 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές πέρασε. 15, τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές περνάει. 18, τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, περνάει. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι πέρασε. 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο παράγραφος 7 υπέρ κατά αποχές περνάει 23 τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές περνάει τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι το ελέγξουμε. Νομίζω ότι πέρασε, αλλά το ελέγξουμε. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει. Περνάει. 28. Υπέρ, κατά. Δεν έχω τις ψηφορίες από το ΕΛ και τους σοσιαλιστές. Για την 28. Α, όλοι κατά. Μάλιστα, αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές περνάει. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε 34 σας παρακαλώ. Άρχεται. Ψετόλοι. Λίγη. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σα... Όχι, λέει πρόεδρος, 41. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, είναι συμβατή, σε ζητώ συγγνώμη. 40. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, περνάει. 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 12. Υπέρ, κατά, αποχές, περνάει. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Όχι, όχι λέει η πρόεδρος. Α, να έρχεται με άλλη μια συμβατή. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά πρέπει να την ελέγξουμε ζητώ συγγνώμη λέει η πρόεδρος τροπολογία 51 άρχεται ψηφοφορία ψηφιστόλη λήξη απορρίπτεται 52. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω το απορρίψετε. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός α. Εδώ έχουμε μια ε, μικρή αλλαγή στη διατύπωση. Νομίζω ότι συμφωνήθηκε να διαγραφεί η λέξεις of approval στην πρώτη τελευταία γραμμή. Vote of approval. Το of approval σβήνει. Λοιπόν, ε, συμβασμός α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται αρχικό κείμενο παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 65, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές. Έχω μπερδευτεί, λέει η πρόεδρος. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 67. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη ψηφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι, λέει η 67. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 69 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Περνάει. «24 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένος 11 ε, υπέρ κατά αποχές ε, περνάει. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές. Φαντάζομαι ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. η ψηφοφορία στην τροπολογία 1. Έληξε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας β, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της αιτιολογικής σκέψης D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές. Φαντάζομαι ότι απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε στην τροπολογία 4 άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Αρχικό κείμενο στο, στην αιτιολογική σκέψη ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του F, του σίγμα τάφ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο του G του Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και άρχεται η ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ε, άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι λίγη ψηφοφορία because he's not with his Okay. Have we finished? Finished? Finished. All right. Have we still got this? Τελειώσαμε. Okay. Thank you very much. That, that finishes the vote. Τελειώσαμε λοιπόν τη ψηφοφορία. Δύο πράγματα ακόμα μας έχουμε να συζητήσουμε. Hang on. Oh, hang on. All right. Oh, sorry to... Well, will somebody give me the list? just a Ναι, ε, ε, προσπαθούμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Here we go. Here we go. Sit down again. Ωραία, ωραία. Καθίστε, για καθίστε. Όσον αφορά ε, την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Ξεκινάμε την τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 και 20 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, τροπολογία 3, υπέρ, Τρία. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 και 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τροπολογία 28 άρχεται ψηφοφορία έληξε Α, με μία φυσικό διαφορά καταπίπτει. Δεν περνάει. 29. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε την 29. Ναι, αλλά άμα δεν σηκώνει τα χέρια σας, τι να κάνω κι εγώ, λέει η πρόεδρος. Άρχεται ψηφοφορία στην 29. Έληξε. Πέρασε. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέρασε. 32 υπέρ. 31. Συγγνώμη, λέει πρόεδρο. Ναι, ναι, μα είναι συμβατή. Το, το λέει και εδώ. Άρα 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Περνάει. 32 υπέρ. Κατά. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 33 και 34 μαζί. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Και θα ήθελα να ελέγξω άρχη την ψηφοφορία. Votes Έληξε. Με μία, ε, μία ακόμα ψήφο κατά, αλλά πέρασε. 37 και 30 35 και 36, συγγνώμη, μαζί. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι περνάει. 37 υπέρ κατά αποχές. Περνάει. 38 υπέρ κατά αποχές. Περνάει. 39 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 41-42 μαζί υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι περνούν. Αλλά να ελέγξουμε τη 41-42 μαζί. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφορία. Ναι, ναι, περνάει. 43 υπέρ, κατά, κατά. αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44-45 μαζί, υπέρ, κατά, κατά. αποχές, εγκρίνεται. 46-47 υπέρ, κατά, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 και 49 μαζί. Favor. Υπέρ, κατά. Κάτα. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά. Αποχές περνάει. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 και 55 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 και 57 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη να, να ελέγξουμε The vote is open on amendment Άρχεται η ψηφορία για τις 56 και 57. Έληξε. Απορρίπτεται. Ε, Εμεί την φωνάξαμε. Τώρα με τι τα χέρια τι να κάνουμε. 58 και 59 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και εδώ. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσατε. Έληξε. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 και 62 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ξέρετε από όταν ψηφίζουν όλες οι ομάδες. 61 και 62. Μαζί. Κλείνει. Απορρίπτεται. 63. Άρχεται. Όχι. Ζητώ συγγνώμη. 63. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Α, κατά πίπτη ναι, ναι. 67 πάμε. Υπέρ, κατά, Λείπουν χέρια από το ΕΛΚ. Ε, μάμα δεν σηκώνει τα χέρια σας. Τι να κάνω. Τι ε, medium είμαι. Υπέρ. 67. Κατά. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Ελέγχουμε. Την 67. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 8. άρχη η ψηφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. 69. Ε, αποσύρθηκε 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι περνάει, αλλά για να το λέξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι λίγοι. Δεν μπορούσα να δω τι κάνουμε. 72. Υπέρ. Κατά. Θα ήθελα να ελέγξουμε την 72. Άρχεται. Έληξε. Περνάει. 73 υπέρ κατά αποχές περνάει. Προφορική τροπολογία στο άρθρο 14. Υπέρ, κατά, αποχές, περνάει. 74 περνάει. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 συνολική τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ Τι είπατε, λέει η Τροπολογία 10. Αποσύρθηκε η χωριστή ψηφοφορία, αλλά εξακολουθούμε να την ψηφίσουμε. 12. Στη 12 είμαστε, τροπολογία 12. Υπέρ, υπέρ τη τροπολογία 12 κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Έληξε. Πέρασε λοιπόν. Σας ευχαριστώ όλους και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Τώρα, Είμαστε στο 17. Εκτό τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στι αναπτυσσόμενε χώρε και στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Περνάει. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ κατά αποχές επαλήθευση τρία έληξε 25 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ξή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, Μα εδώ ψηφίζουν μερικοί και τις δύο Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα ξανά υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίθηκε. Εφτά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 με προφορική τροποποίηση. Την όλοι υπέρ, κατά, αποχές. Θα επαληθεύσουμε την, την 14, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, έληξε. 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 15 σε δύο τμήματα. Ένα, πρότεινα ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Α, όχι, τώρα υπάρχει μια σειρά 23, 24 και 25 μαζί. Υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνονται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν απέχουν οι σοσιαλιστές εγκρίνεται 30 υπέρ είναι προφορική. Είναι με προφορική υπέρ λοιπόν. Δεν είναι σε τιμήματα. Είναι προφορική τροποποίηση ώστε να διαγραφεί το including illegal immigration. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η φράση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 εγκρίνεται νομίζω 40 υπέρ κατά όχι. εγκρίνεται 41 υπέρ κατά όχι. εγκρίνεται έχει καταπέσει 42 43 υπέρ κατά όχι. εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. «37 υπέρ 2 αποχές». Ορίστε, τελείωσε. Σας υπενθυμίζω ότι το απόγευμα θα είμαστε στο ημικύκλιο για την ακρόαση, για την εποπτεία. Στο ημικύκλιο. Ευχαριστώ πολύ.